Το σύμφωνο αυτό πάντως θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε απειλή για την ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Σικέρσκη. Λίγη εδώ αυτό το τμήμα. Είχαμε και την κυρία Ματέρα στον κατάλογο για τις μονόλεπτες, αλλά επειδή απουσίαζε δεν έλαβε και το λόγο. Γι' αυτό έληξαν εδώ οι μονόλεπτες παρεμβάσεις. Κάποιε από αυτέ τις παρεμβάσεις κράτησαν πάνω, πολύ πάνω από ένα λεπτό, δύο λεπτά. Συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη έκθεση Σάντεμο για την γενική ασφάλεια προϊόντων και την εποπτεία στην αγορά. Η κυρία εισηγήτρια έχει τον λόγο. Έχετε τον λόγο κυρία εισηγήτρια. Γνωρίζοντας βέβαια ότι έχετε τέσσερα λεπτά φυσικά και θα έχετε μπορείτε να φτάσετε έως τα 6 λεπτά. 4 συν 2 για την εισηγήτρια. Σωστό. Έχει τον λόγο η κυρία Σαντεμόζο. Τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα. Σύντομα θα σας αναφέρω Περί τίνος πρόκειται σε αυτή την έκθεση που προετοιμάστηκε από την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών. Είναι μια έκθεση για την αναθεώρηση τη οδηγία για τη γενική ασφάλεια και την εποπτεία στι αγορέ πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία και την προετοιμάσαμε επειδή σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να αναθεωρήσει την ε, οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Πράγμα που σημαίνει για μα μια καλή δικαιολογία κατάθεση έκθεση που αναφέρεται σε αυτή την αναθεώρηση τη οδηγία για τη γενική ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Διαιρέσαμε σε δύο την δομή αυτή τη έκθεση χωρίσαμε σε δύο τμήματα. Υποβάλλουμε κάποιε συστάσει για το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την εποπτεία τη της αγορά γενικά και πιο συγκεκριμένα, πιο εξειδικευμένα, έχουμε πιο εξειδικευμένε συστάσει για την αναθεώρηση του περιεχομένου τη οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Πρώτα απ' όλα, όταν πριν από κάποια χρόνια εγκρίθηκε η οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων, μετατράπηκε σε ένα ορόσημο όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και εξακολουθεί να είναι ορόσημο. Όμως έχουμε κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή, διότι στην πραγματικότητα η εποπτεία της αγοράς δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όπως επιθυμούσαμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές θα είναι επαρκώς ασφαλείς. Γι' αυτό στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή προτείναμε να γίνει μια προσπάθεια διπλή προσπάθεια ώστε να ε, προσαρμοστεί η εποπτεία στην αγορά. Σε μια περίοδο κρίσεως υπάρχει ο κίνδυνος στα κράτη-μέλη να μην δώσουν περισσότερους πόρους στην εποπτεία της αγοράς, αλλά λιγότερα κονδύλια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις, που είναι εκείνες που πρέπει να ανταποκριθούν στις ρήτρε και διατάξεις που ισχύουν στην εσωτερική αγορά. Προετοιμάζοντα αυτή την έκθεση, συζήτησα με πολλέ επιχειρήσει που δρούν στην εσωτερική αγορά και πολλέ αυτέ τι επιχειρήσει μου λένε ότι ποτέ ποτέ δεν υπήρξαν αντικείμενο κάποιου ελέγχου ή κάποιου μέτρου εποπτείας ή επιτήρησης της αγοράς σε σχέση και με αυτό που δημιουργεί ακριβώς και προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν υπάρχουν αξιολογήσεις και τίση έλεγχοι, τι γίνεται τουλάχιστον υπάρχει, για να υπάρχει ένας ισότιμος ανταγωνισμός και να τηρούνται οι διατάξεις και τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν σαφώς στην εσωτερική αγορά με το σωστό τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για τις επιχειρήσεις να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο στην αγορά για αυτά τα θέματα. Θα περάσω σε κάποια από τα πιο εξειδικευμένα μέτρα που προτείνουμε για την αναθεώρηση τη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Είναι σαφέ ότι η πλειοψηφία των προτάσεων που κάνουμε είναι προ όφελο των καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθεί η ίχνηλασιμότητα, η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων προϊόντων στην αλυσίδα είναι θεμελιώδου σημασία αν θέλουμε να αποσύρουμε από την αγορά κάποια επικίνδυνα προϊόντα. Επίση, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να δρουν γοργά όταν ανοιχνεύεται η ύπαρξη επικίνδυνων προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ προϊόντα που εισέρχονται από τρίτε χώρε, χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερο εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα από αυτέ τι χώρε στην Ευρωπαϊκή Αγορά και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκρίνονται στι διατάξει που ισχύουν για τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά που παράγονται από τα δικά μα κράτη. Θέλουμε να είναι πιο εξειδικευμένη η νομοθεσία και γι' αυτό στην έκθεσή μα προτείνουμε επίση να υπάρξει στατιστική υποχρεωτική στατιστική για τα συμβάντα, τα ατυχήματα, να γνωρίζουμε επαρκώ σε ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα σε σχέση με τα ατυχήματα και τα συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί, έχουν ανακύψει προηγούμενα. Έτσι μπορούμε να εξειδικεύσουμε το νομοθετικό μα έργο και να το στοχοθετήσουμε επικεντρωνόμενοι στου πιο αναγκαίου τομεί, χωρί να στρεβλώνονται ή να δημιουργούνται προβλήματα για του ασφαλεί τομεί και ασφαλή προϊόντα. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνεται στα προϊόντα στην, που πολλούν σε ε, γραμμή, σε αλυσίδες, διότι πολλές φορές υπάρχουν παράπονα ότι δεν υλοποιούν πάντα τις ρήτρες και τις διατάξεις ασφάλειας, όπως τα προϊόντα που αγοράζονται σε μαγαζιά, αυτά τα οποία πολλούνται για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, online, σε, στη γραμμή, ηλεκτρονική γραμμή εννοείται και να δούμε και τι μπορεί να γίνει για την ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα να είχαμε δώσει μεγαλύτερη προσοχή πώς θα προστατεύαμε τα παιδιά, τους ανήλικους. Δυστυχώς όμως ε, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς δεν ε, ήταν δυνατό να επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία για ειδικέ ρήτρε που πρέπει να λειτουργήσουν υπέρ των παιδιών αλλά και πιο εξειδικευμένα μέτρα υπέρ των ανήλικων. Θέλω να πω λοιπόν ότι θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων. Είναι σαφές αυτό αναγκαίο να ενισχυθεί η εποπτεία των αγορών και είναι αναγκαίο η εποπτεία αυτή να είναι συνεκτική και με συνεκτικότητα ώστε να λαμβάνονται υπόψη εκείνα τα μέτρα νομοθετικά τα οποία χρειάζονται και να είμαστε αποτελεσματικοί ώστε να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές στην ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζουν και οι επιχειρήσεις να έχουν ένα ισότιμο πλαίσιο για τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Με αυτά ολοκλήρωσα. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δυνατόν γοργότερα να υλοποιήσει αυτή την αναθεώρηση σε σχέση με αυτή την οδηγία και από τα κράτη-μέλη να δώσουν επαρκή κονδύλια για να διασφαλιστεί η εποπτεία τη αγοράς όπως οφείλουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τον γύρο Catch the Eye. Η κυρία εισηγήτρια κατανάλωσε τον χρόνο που είχε στη διάθεσή τη ε, ούτω ή άλλω και θα ακούσουμε τώρα του συναδέλφου που ζήτησαν τον λόγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα λάβει τον λόγο πρώτα η κυρία Λάρα Κόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαίρω την ε, συνάδελφο, την κυρία Σάλντε Μόζε, για την επικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε. Ήθελα να δώσω έμφαση στο εξή. Στην έκθεση της Επιτροπής ΙΤΕ, πολύ σωστά αναφέρεται το εξή στοιχείο που και εμεί θέλαμε και ευχαριστώ την κυρία Σάλντερ ε, γι' αυτό. Ότι θα χρησιμοποιήσουμε και τα νέα τεχνολογικά μέσα όπω τα μικροτσίπ ή οι ραδιοσυχνότητε, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο εντοπισμό, εντοπισμό των προϊόντων. Έτσι εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των ε, καταναλωτών και καλύτερη ποιότητα για τα προϊόντα. Επίση, καλύτερη ίχνηλασιμότητα των προϊόντων, ώστε ο καταναλωτή να είναι σε θέση να γνωρίζει όλε τι πτυχέ που αφορούν το προϊόν τι διάφορε φάσει κατασκευή του, την προέλευση των ε, πρώτων υλών και το ποιοι είναι υπεύθυνοι για το κάθε στάδιο παραγωγής. Επίσης δεν θα χρειάζεται πλέον το κριτήριο τη ε, ε, κατάδειξη τη προέλευση ενό προϊόντο με το Made in. γι' αυτό για ένα προϊόν που λέγεται χαρακτηρίζεται ως made in France ενώ εκεί γίνεται μόνο συναρμολόγηση λόγω χάρη του προϊόντος, αυτό είναι παραπλανητικό στοιχείο για τον, καταναλωτή. Έτσι ελπίζουμε ότι η Επίτροπος θα λάβει υπόψη την αίτηση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να έχουν καλύτερη ε, ενημέρωση όλοι οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι έχετε αυστηρά ένα λεπτό για τις παρεμβάσεις σας, αγορητές. Η κυρία Τικάου τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τη συνάδελφο για αυτή την έκθεση. Την ευχαριστώ επειδή δέχτηκε και τη δική μας την τροπολογία στην ψηφοφορία της Επιτροπής ΙΤΡΕ και να θυμίσω εδώ τη σημασία των ευρωπαϊκών προτύπων και για τους διαγωνισμούς που οργανώνονται είτε είναι κλασικού τύπου είτε ηλεκτρονικοί σε κάθε περίπτωση αυτό μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε του καταναλωτέ ώστε να έχουμε καλύτερη ασφάλεια των προϊόντων. Μα ενδιαφέρει επίση να ακολουθούνται αυστηρά οι διαδικασίε τυποποίηση, ακόμα και στι ιδιωτικέ σχέσει και στα πολιετή προγράμματα. Θέλουμε το όλο σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά. Επίση, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονό ότι χρειάζεται απλούστευση των ευρωπαϊκών προτύπων και η σύνταξή τους να γίνει πιο αποτελεσματική. Θα θέλαμε λοιπόν οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης να μειώσουν το χρόνο επεξεργασίας του κάθε προτύπου. Η κυρία Φιγκερέδο θα λάβει τώρα τον λόγο παρακάτω. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει τεράστια σημασία να δώσουμε την προσοχή μας όπως πρέπει στις ρήτρες ασφάλειας των προϊόντων με μια προοπτική όχι μόνο προάσπισης ε, της παραγωγής αλλά επίσης και προάσπισης των καταναλωτών εξίσου. Η απλούστευση των διατάξεων και των προθεσμιών δεν μπορεί να υπονομεύει τα εχέγγυα που χρειάζονται και πρέπει να έχουν οι καταναλωτές μας. Και επίσης όταν βλέπουμε και στρέφουμε την πτυχή μας για αυτές τις πτυχές, αυτές τις πτυχές ασφάλειας δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα προϊόντα τα οποία εισάγουμε και εξίσου την προάσπιση της ένδειξης που έχει παραχθεί στην Made in που είναι πάρα πολύ σημαντική ένδειξη και γι' αυτό αναμένουμε να λάβει υπόψη αυτές τις πτυχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπεριέχονται σε αυτή την έκθεση τις παρεμβάσεις που επίσης η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου έκανε για την εξειδίκευση των προτάσεων και που έγιναν δεκτές από την εισηγήτρια και έτσι θα μπορέσουμε στο τέλος τέλος να προχωρήσουμε κάπως παραπάνω στην προάσπιση της ασφάλειας των προϊόντων των παραγωγών και των καταναλωτών εξίσου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φίγερ εδώ. Τώρα ο κύριος Όμπερμαϊερ παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην έκθεση γίνεται λόγο για μεγάλε λέει προόδου. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε ω επιφύλαξη ότι παρόλα αυτά για την οδηγία, για τα παιχνίδια και παρότι υπάρχουν αυτέ οι προσπάθειε, 60 περίπου 100 των προϊόντων προέρχονται από την Κίνα. Και το μεγαλύτερο μέρο των επικίνδυνων αυτών προϊόντων προέρχονται από μια αγορά που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι το νέο σύστημα που θα δημιουργηθεί θα ανακουφίσει αυτή την κατάσταση. Πρέπει με σθένο να υιοθετήσει μια θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει την υγεία και την προστασία των καταναλωτών. Ιδιαίτερα μα εκπλήσει ότι ένα τέταρτο των προϊόντων που είναι παιχνίδια, πιστόλια και άλλα τέτοια θέσει ε, παιδιών, ε, θέσει ε, καθίσματα για τα παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω αντιδρά πολύ αργά σε αυτά τα προϊόντα. Και έτσι βλέπουμε σε σχέση με την παραγωγή κάποιων υπάρχουν απαγορεύσεις. Ωστόσο όμω ήταν γνωστή η επιζήμια, οι επιζήμιες αυτές Καταστάσει που προκαλούνται για την υγεία αυτών των παιδιών εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Και υπάρχουν τέτοια παιχνίδια και προϊόντα που δεν έχουν απαγορευτεί. Πρέπει η ανάκληση αυτών των προϊόντων πιο γοργά και πιο αποτελεσματικά να διαμορφώνεται στην αλυσίδα των ε, πολιτών, ώστε να είμαστε πιο ε, αποτελεσματικοί. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτοβα τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εδώ και καιρό ψάχνουμε να βρούμε μέτρα που να επιτρέπουν καλύτερη λήψη υπόψη όλων των συμφερόντων των ενδιαφερομένων στην εσωτερική αγορά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός, να προβλεφθούν ποινικέ κυρώσεις δε. Επίσης, υποστηρίζω την υποχρεωτική δημοσίευση των αξιολογήσεων πριν δοθεί οποιοδήποτε δάνειο διότι τα επικίνδυνα προϊόντα συχνά προέρχονται από τρίτες χώρες και γι' αυτό είναι ουσιώδες την υποχρέωση αυτή να τη συμπεριλάβουμε όχι μόνο για Ευρωπαίους αλλά και για διεθνείς παράγοντες και στις διεθνείς συμφωνίες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρόικοβα. Σας ευχαριστώ. Βεσλούνται και ολοκληρώνεται αυτός ο γύρος παρεμβάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαντεμόζε για μια εξαιρετική έκθεση. Για άλλη μια φορά θέλω να υπογραμμίσω το γεγονό ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια και πρέπει να είμαστε πιο εξειδικευμένοι για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων. Ω καταναλωτέ διαβάζουμε δημοσιεύματα στον τύπο επανειλημμένα και μαθαίνουμε σε σχέση με οργανώσει προστασία καταναλωτών που κάνουν δοκιμασίε, κάνουν τέτοια τεστ και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πράγματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και που μπορούν να είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα, μοιραία ίσως κιόλα και για τα παιδιά. Και ε, τα προϊόντα αυτά που θεωρούνται ασφαλή δεν είναι ασφαλή. Είναι, το πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα των χημικών που περιέχονται. Πολλά τέτοια προϊόντα έχουν χημικέ ουσίε που ήδη απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω χρησιμοποιούνται ακόμα. Και είναι πολύ δύσκολο οι επιμέρου καταναλωτέ να κατανοήσουν και να δουν τι πρόβλημα υπάρχει με αυτά τα προϊόντα. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση, να συντονιστούν μεταξύ του ώστε να απαγορευτούν αυτά τα προϊόντα από την αγορά πρέπει να πείσουμε του παραγωγού να μην θέτουν σε κυκλοφορία τέτοιου είδου προϊόντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ακούγοντα την Επίτροπο, κυρία Δαμανάκη που σίγουρα ευχαριστώ οπωσδήποτε για την παρουσία της εδώ αυτή την ώρα και την προσοχή με την οποία παρακολούθησε αυτή τη συζήτηση όχι μόνο όπω ήταν η υποχρέωσή της αλλά και τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού που έγιναν στον προηγούμενο γύρο. Κυρία Δαμανάκη έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you, President. It... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί βλέπουμε από όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως γυναίκες, να συμμετέχουν ε, σε όλο αυτό το θέμα. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Εδώ λοιπόν να συγχαρώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ευρωκοινοβούλιο για το ψήφισμα που ετοίμασε για την αναθεώρηση της οδηγίας για την κοινική ασφάλεια των προϊόντων και υποπτία της αγοράς. Να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει αυτή την έκθεση και εκτιμά την ποιότητα, την πολύ καλή ποιότητα του περιεχομένου. Ε, τα πορίσματα της έκθεσης αυτής ε, συμπίπτουν ε, με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ να αναθεωρήσει τι ε, προδιαγραφέ για τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα σαφέ ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό μαζί σα. Ένα πλαίσιο που να, να προσδίδει ένα εσωτερικό σύστημα ε, καλή και ασφαλού κυκλοφορία των προϊόντων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξαγάγει ευρείε διαβουλεύσει με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να ορίσει πώ θα πετύχουμε αυτό το στόχο για να έχουμε μια συνεκτική λύση μεταξύ όλων των διαφόρων τομέων προϊόντων, ο αντιπρόεδρο Ταγιάννη και ο επίτροπο Ντάλι συμφώνησαν να συνεργαστούν προκειμένου να πετύχουν αυτή την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων για την εποπτεία τη Ευρωπαϊκή Αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διαβεβαιώσει ότι και να εξασφαλίσει μάλλον ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα υποφελούνται από προϊόντα καλής ποιότητας. Πρέπει έτσι λοιπόν να αναθεωρήσουμε τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς κανόνες για τα προϊόντα, ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να λάβουμε μέρημνα και του περιθωρίου ελιγμών που διαθέτουμε βεβαίω και να σεβαστούμε και τι αρμοδιότητε των εθνικών κρατών μελών, όπω τα καταλαβαίνετε και μόνοι σα. Ωστόσο, οι κανόνες θα μπορούν να μας, θα μας επιτρέψουν να εντοπίζουμε εύκολα και να αντιμετωπίζουμε κατεπίγουσες ανάγκες νέων κινδύνων. Συμφωνώ ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι στην νέα λυσίδα κυκλοφορία των προϊόντων. Συμφωνώ επίση ότι η προστασία των παιδιών, η μερέγγιμα των παιδιών είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Ε, ταυτόχρονα η αναθεώρηση θα πρέπει να δώσει ισότιμους και ισοδύναμους κανόνες για όλους τους ε, συμμετέχοντες ε, και συνελασσόμενους στην αγορά, ε, ιδίω για, για το διοικητικό κόστο. Θα πρέπει επίση να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των κανόνων για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπω το ορίζει η σχετική οδηγία, και τους κανόνες του πακέτου του 2008 για τα προϊόντα. Αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Προφανώς οι υποχρεώσεις για την ασφάλεια ενός προϊόντος θα πρέπει να καθορίζονται για τους ε, οικονομικούς φορείς. Και εδώ χρειάζεται συντονισμός ε, και καλύτερη εποπτεία της ε, αγοράς των κρατών μελών. Τέλος, το να λειτουργήσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα προϊόντα που δεν προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση, το RAPEX, είναι κάτι που θα είναι καθοριστική σημασία. Αυτό ήδη το έχουμε χρησιμοποιήσει για τη συνεργασία μα με την Κίνα και άλλε χώρε. Συμφωνούμε λοιπόν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί αυτό το σύστημα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα απειλών που εδώ αναφέρονται. Ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη και ο Επίτροπος Ντάλι σκοπεύουν από κοινού να υποβάλουν μια πρόταση για, μια για ένα ενιαίο και συνεπές ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς. Σας ευχαριστώ ξανά για αυτό, την πολύ καλή... για αυτό το πολύ καλό ψήφισμα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίματων. Ψηφίσματος θα γίνει αύριο το μεσημέρι, 12.00. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη.